Sehr Αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε στις ε, επεξηγήσεις ψήφου και θα ήθελα όλοι σας να φύγετε και να ακούσουμε αυτούς οι οποίοι πρέπει να λάβουν το λόγο ή που θέλουν ακόμα να λάβουν το λόγο. Παρακαλώ αποχωρήστε ταχαίως ώστε να μπορέσουν να ομιλήσουν οι επεξηγούμενη